Καλημέρα σας. Ψηφίζουμε äh, την έκθεση του συναδέλφου Φίσας για την ευρωπαϊκή γαστρομική κληρονομιά, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές. Θέλει να πει τίποτα ο εισηγητής, παρακαλώ κύριε Φίσας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ Ντόρις αγαπητή. Ε, πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες, όλους τους κοιόδης ηγητές για τη συνεργασία τους στην έκθεση αυτή. Εγκρίθηκε η μεγάλη ε, πλειονότητα των τροπολογιών, έγιναν πολλοί συμβασμοί και με στόχο την ομοφωνία το θέμα είναι πιο σημαντικό από ό,τι φαίνεται ενδεχομένω εκ πρώτη όψεω. Έχει να κάνει και με την υγεία των νέων μα στο μέλλον, αλλά και την προστασία μια τόσο σημαντική πολιτιστική κληρονομιά που είναι η γαστρονομία. Για όλη την Ευρώπη είναι και πηγή απασχόληση εξάλλου και πλούτου και τουρισμού. Γνωρίζω ότι οι φιλελεύθεροι έχουν άλλη άποψη, αλλά του ευχαριστώ παρόλα αυτά που την κατέθεσα. Υπάρχουν και κάποιες ε, προφορικές ε, τροπολογίες, ε, δεν χρειάζεται να τις διαβάζουμε στη συνέχεια, βέβαια η Πρόεδρο θα αποφασίσει, διότι έχουν κυκλοφορήσει, είναι υπόψη όλων των πολιτικών ομάδων και συμφωνούν. Επαναλαμβάνω λοιπόν τι ευχαριστήσει μου και προς τους βοηθούσε την δική μου συνεργάτη Μαρία Φουνιέ και όλους τους υπολείπους που εργάστηκαν προς την κατεύθυνση αυτή για να έρθει το κείμενο σε ασιοπέρας και με πολύ μεγάλη ε, συμφωνία. Ευχαριστώ. Αρχίζουμε λοιπόν. Συμβαστική εναίπε, κατά αποχέ εγκρίνεται. Η τροπολογία 46 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 52 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. 53 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 54 είπε. Καταπίπτει. Ζητώ συγγνώμη. 55. επε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 είπε κατά αποχές απορρίπτεται 57 είπε κατά αποχές εγκρίνεται 58 είπε κατά αποχές εγκρίνεται 59 έχει αποσυρθεί 60 είπε κατά αποχές εγκρίνεται 61 είπε κατά αποχές εγκρίνεται η συμβιβαστική 3 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Η ε, συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το πρώτο τμήμα ήταν αυτό, δεύτερο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 72 ε, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ, κατά, ξανά παρακαλώ υπέρ, κατά αποχές. Δεν χρειάζεται έλεγχο γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εντάξει, εντάξει, ναι, σα μετράω. Πέρασε. Ένα 16 εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 77. Υπέρ. 74, συγγνώμη. 70... Ε, Τρέχω, 74 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. 75 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται. 76 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 77 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 79 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 80 σε δύο τμήματα τρίμα πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100. Υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχη ψηφοφορία. Τροπολογία 100.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 108 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ, όχι, έχει αποσυρθεί. 111 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά αποχές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 αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία. closed. Πέρασε.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 κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία πρώτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία αρχίζει Πέρας. Δεκαεννέα ψήφι υπέρ, χωρίς αποχές, χωρίς ψήφους κατά και συγχαρητήρια. Κύριε Φίσας, καλή ιδέα λοιπόν είχατε. Δεν πίστεψαν όλοι ότι θα στεφθεί με επιτυχία. Χωρίς μικρόφωνο. Χαίρομαι που συμφωνεί στο τέλος. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε στον κύριο Λόκεχαρτ, ο οποίος δεν μπόρεσε να προσέλθει σήμερα. Είναι όμως τεχνική τύπου μόνο ψηφορία. Και αρχίζουμε. Τροπολογία πρώτη, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική. Μία και δύο υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελευταία, τελευταία ψηφοφορία, τελική ψηφοφορία. Αρχίζει. Δεκαεννέα επέρ, μία ψήφος κατά εγκρίνεται. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες και τώρα θα περιμένουμε να έρθει η κυρία Ρέντινγκ. Η Επίτροπος Παρακαλώ μη φύγετε όλοι. Μη με αφήσετε μόνη μου. Θα είναι μεγάλος ο αγώνας, μεγάλη μάχη. Καλύτερα να είσαστε κοντά μου. Για τη Ρέντινγκ την ίδια.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 begrüße, möchte ich gerne... Καλημέρα σας. Θα ήθελα να καλωσορίσω την ε, Επίτροπο. Έχουμε και μια ομάδα επισκεπτών από την Αυστραλία. Έρχονται σε αυτή την ψύχρα που έχουμε εμείς από πολύ ζεστά κλίματα. Μακάρι να είχαμε να σας δείξουμε και λίγο χιονάκι, αλλά δεν τα καταφέραμε. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπουμε εδώ λοιπόν. Έχετε την τακτική σας συνεδρίαση ε, με την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. Σας έφερε εδώ ο κύριος Τάκουλα, ο συνάδελφος. Σήμερα το πρωί θα παρακολουθήσετε, φαντάζομαι με χαρά, την ε, Επίτροπο και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε συζήτηση μαζί της. γιατί θα μας παρουσιάσει τα θέματα τα οποία έχει ολοκληρώσει κατά την ε, θητεία της και άλλα ζητήματα τα οποία ακόμη σας δεν έχουν προχωρήσει επιτυχώς. Αγαπητή Βιβιάν Ρέντινγκ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ένα θερμό καλώς όρισμα και προς τους προσκεκλημένους ε, μας. Θα ήθελα να πω στους βουλευτές με τους οποίους εδώ και 15 χρόνια συνεργαζόμαστε σε αυτή την Επιτροπή. Πώς έχουμε εκλογές σε ακριβώς 100 ημέρες, όχι χρόνια, όπως μου ξέφυγε και είπα, θα είμαστε σε πλήρη αναβρασμό. Και θα είναι πολύ διαφορετικές οι εκλογές αυτές από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Θα είναι πραγματικά μια εκλογική αναμέτρηση αυτή η οποία θα ορίσει το είδος της Ευρώπης που θέλουμε στην οποία θέλουμε να ζούμε. Και γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να είναι ενήμερος ο ψηφοφόρος για τις πολύ σημαντικές αποφάσεις που έχει να λάβει. Μαζί σας λοιπόν θα ήθελα να κοιτάξω εν συντομία τα επιτεύγματά μας Τώρα στις αρχές του 2014 μπορούμε να στρέψουμε το βλέμμα προς τα, το βλέμμα προς τα πίσω, κάποια χρόνια. Η ευρωπαϊκή ηθαγένεια, η προσέγγιση δηλαδή με τόσους πολλούς ε, πολίτες έχει, έχει στεφτεί με επιτυχία. Ο διάλογος με τον πολίτη έχει αναπτυχθεί σε 15 τουλάχιστον περιπτώσεις με διαφόρους επιτρόπους και εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πολλά κράτη-μέλη και με πολλούς ε, υπουργούς εθνικών κυβερνήσεων στο διάλογο αυτό με τους πολίτες. Είχαμε παρουσία και πολλών χιλιάδων πολιτών μέσα στις αίθουσες των συνομιλιών αλλά και πολλών άλλων ε, παρουσία όχι ε, πραγματική αλλά πλασματική μέσω του διαδικτύου και των παρατηρήσεων που μας έστελαν από το Facebook και το Twitter. Και εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι επιτροποί έχουμε επίσης αναπτύξει διαδικτυακούς, διαγραμμικούς διαλόγους. Επικοινωνία κυρίως με τους ιστολόγους. Αυτοί οι διάλογοι ιστολογικοί έχουν μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τους παρακολουθούν κυρίως οι νεότερες γενναίες μέσα από το διαδίκτυο και συνεχίζουμε τους διαλόγους αυτούς. Στην αρχή της εβδομάδας βρισκόμουν στο Λονδίνο μάλιστα. Σε δέκα μέρες θα είμαι στη Βαρκελόνη, λίγο μετά ο Επίτροπος Μπαρνιέ στο Παρίσι. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την επικοινωνία για να αναπτύξουμε έναν πανευρωπαϊκό διάλογο και εδώ στις Βρυξέλλες, όπου θα έχουμε προσκεκλημένους ε, από τις 50 ε, αυτές εκδηλώσεις των διαλόγων και βέβαια και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι βουλευτέ είναι προσκεκλημένοι να έρθουν στον πανευρωπαϊκό, στο μεγάλο διάλογο, για να ολοκληρωθεί πριν από τι εκλογέ, γιατί βεβαίω δεν θέλουμε καμία παρεμβολή στην εκλογική εκστρατεία. Θέλουμε να αφήσουμε το χρόνο και σε εσά να προετοιμάσετε τι εκλο... προεκλογικέ εκστρατείε. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μαζί και με εσά αναπτύξει νέε πρωτοβουλίε, τι έχουμε θέσει σε λειτουργία Έχουμε παραδείγματι για τρίτη χρονιά το Share Europe Online. Καταρτίζουμε στα γραφεία ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσωπικό υπαλλήλου, ώστε να είναι σε θέση αυτοί να απευθύνονται στο κοινό, στον πολίτη και μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Ήταν μια ε, ιδέα της Μαρίτσα Σάκ και του Νόρτεν Ντοχτέρπατ. Πολύ καλή ιδέα πρέπει να συνεχιστεί. Επίσης έχουμε το New Narrative for Europe, ε, νέα, νέες επιλογές, επιλογές για την Ευρώπη με επιστημονικό ε, ιδιαίτερα προσωπικό, όπου με την Επίτροπο Βασιλείου και τον κύριο Μπαρνιέ αναπτύξαμε προσωπικά την ε, πορεία αυτή για να προσεγγίσουμε την Ευρώπη που δεν έχει οικονομική τόσο βαρύτητα αλλά έχει μεγάλη πολιτιστική και επιστημονική αξία με αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν σε επόμενους μήνες. Για πρώτη χρονιά επίσης λειτουργεί ένα άλλο πιλωτικό σχέδιο Promise for Europe υπόσχεση για την Ευρώπη. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ε, προσέγγιση προς όλες τις γενιές στην Ευρώπη για να δούμε τα κοινά οράματα, την κοινή αντίληψη για την Ευρώπη και θα κάνουμε τη χαρτογράφηση αυτών των προσεγγίσεων του τι είναι Ευρώπη σε, για να σημειώσουμε σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει η αντίληψη στο κάθε κράτος μέρος από τα δέκα που έχουν επιλεγεί. Μια νέα επιχειρησιακή προσέγγιση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση που σημαίνει ότι εργαζόμαστε διοργανικά για να αναπτύξουμε ένα ενιαίο συλλογικό μήνυμα και όχι ένα συνονθήλευμα αντιφατικών μηνυμάτων. Με την ιδέα ότι κοιτάμε το δάσος και όχι τα δέντρα δηλαδή. Αυτό το έχουμε ήδη ξεκινήσει και ενισχύουμε έτσι την αποτελεσματικότητα της επικοινωνιακής μας πολιτικής. Επίσης, σε μια τελική επιτάχυνση ενόψη των εκλογών τον Μάιο, συνεργαζόμαστε και έχουμε υπογράψει ε, μνημόνιο συνεννόησης για τα 500 κέντρα άμεσης πληροφόρησης, ώστε η Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο για τις δραστηριότητες του Europe Direct και από πλευρά σας η Επιτροπή του Πολιτισμού να μας υποδεικνύει σε πρώιμο στάδιο το πώς θέλει το, το, δίκτυο των κέντρων πληροφόρησης του Europe Direct να συμμετάσχει και να συμβάλλει στην προεκλογική σας εκστρατεία. Ήδη εκπαιδεύεται το προσωπικό των κέντρων αυτών πληροφόρησης για να είναι σε θέση να στηρίξουν με την τεχνογνωσία τους ε, και την εργασία τους τους υποψηφίους. Έχουμε σε αυτό συνεργαστεί με τους δύο αντιπροέδρους σας, Άννη Ποντιματά και Ότμαρ Κάρας, για μια ε, ενισχυμένη διοργανική σε επίπεδο δηλαδή συνεργασία. Έχουμε, απευθύνει, έχουμε καταγράψει επιστολή τους κοινού μας στόχους. που απευθύνεται στις ε, στα γραφεία πληροφόρηση του Κοινοβουλίου και τη Αντιπροσωπή τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό για να υπάρχει μια κοινή ε, στάση, να δουλεύουμε όλοι μαζί ως ομάδα. Αλλά ξέρετε βέβαια τι πρόκειται να συμβεί με τις εκλογές, όπως πάντα οι ευρωεκλογέ θα έχουν και τοπικό χρώμα, γι' αυτό και θα πρέπει να ακούσουμε και τι συστάσει των εκπροσώπων μα στα ε, ε, κατατόπους γραφεία ώστε να αναπτυχθεί η εκστρατεία κατά τρόπο διαφορετικό. Φαντάζομαι στη Φιλανδία από ό,τι στην Ισπανία ή από το Λουξεμβούργο στην Ουγγαρία. Δεν θα είναι το ίδιο πράγμα πάντα. Πρέπει να ακούσουμε δηλαδή τι έχουν να μας προσφέρουν με τις γνώσεις τους για την κατατόπους κατάσταση οι εκπρόσωποι μας εκεί. Το Europe Round the Corner επίσης είναι μια ιδέα που έχει ξεκινήσει από την αντιπροσωπεία μας στις κάτω χώρες, η Ευρώπη της διπλανής πόρτας, θα εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη με ε, διαγραμμικαίους πόρους που θα εξασφαλίσουν ε, την συλλογή όλων των χρηματοδοτικών πόρων σε ένα μόνο πακέτο θα μπορείτε, ε, στο οποίο θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση εσείς στην εκστρατεία σας ώστε να γνωρίζετε τι μπορείτε να αξιοποιήσετε σε τοπικό επίπεδο από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έτσι αντιμετωπίζεται ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, διότι ο πολίτη πολύ συχνά δεν γνωρίζει τι είδους έργο χρηματοδοτείται στην περιοχή του από ευρωπαϊκά κονδύλια και έτσι θα μπορείτε εσείς να βλέπετε κατά την εκστραστία σας μέσω του εργαλείου αυτού τι είδους χρηματοδότηση προβλέπετε στην κάθε περιοχή για να ενημερώνετε τους πολίτες για τις επενδύσεις που έχουν γίνει στον τόπο τους. Επίσης, ε, περιθυμίζω τις συστάσεις της Επιτροπής να υπάρχει ένας εκπρόσωπος από κάθε πολιτική οικογένεια για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα ψηφοδέλτια να καταγράφουν ποια είναι τα εθνικά κόμματα τα οποία ανήκουν στην συγκεκριμένη αυτή πολιτική οικογένεια, στο Ευρωπαϊκό Κόμμα δηλαδή. Να έχουμε δηλαδή τον παραλληλισμό, την, την καταγραφή του ευρωπαϊκού και, του εθνικού, και των εθνικών κομμάτων μαζί. Αυτό είναι κάτι πρέπει να κάνουμε σε δύο επίπεδα, και, στο ευρωπαϊ, και ευρωπαϊκά και στα εθνικά κόμματα. Από την τελευταία μας έκθεση επίσης είχαμε δηλώσει ότι θα, θα... θα αναπτύξουμε ένα εγχειρίδιο των δικαιωμάτων των πολιτών, ένα απλό κείμενο, φυλάδιο, το οποίο θα εξηγεί στον πολίτη με απλούς όρους τα δικαιώματα που έχει. Θα δημοσιευθεί και αυτό και θα διαδοθεί, θα διατεθεί μέσα στους προσεχείς μήνες και βέβαια πριν από τις ευρωεκλογέ. Και αγαπητοί συνάλφοι, δεν θα μπορούσα βέβαια να προσέλθω στην Επιτροπή σας χωρίς να μπορώ να, χωρίς να είμαι έτοιμη να σας πω για τα τελευταία αυτά 15 χρόνια που είμαι επίτροπος και που πάντοτε είχα ιδιαίτερο σύνδεσμο με την Επιτροπή του Πολιτισμού, γιατί στην πρώτη μου θητεία είχα την αρμοδιότητα εκπαίδευση και του πολιτισμού, μετά τη κοινωνία των πληροφοριών και των ασφαλιστικής ενημέρωση και τώρα τη Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Και με αυτό το τίτλο βρίσκομαι πάλι ενώπιον σα. Η Ιθαγένεια λοιπόν, όταν πριν από 15 χρόνια ξεκίνησα, ήταν μια θεωρία επιχάρτου. Και νομίζω ότι πια την ε, αναπτύξαμε, της δώσαμε φτερά και αντιλαμβάνεται πια ο πολίτης ότι δεν είναι μόνο ο πολίτης μιας περιοχής, μιας χώρας, αλλά και ότι είναι και πολίτης της Ευρώπης. Πράγμα το οποίο αποδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις μας από το Ευρωβαρόμετρο, διότι ο πολίτης από ό,τι φαίνεται γνωρίζει ότι είναι πολίτης της Ευρώπης. Δεν ξέρει ακριβώς τι σημαίνει πάντα το ότι είναι πολίτης της Ευρώπης, αλλά ξέρει ότι είναι πολίτης της Ευρώπης. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω κάποια από τα ορόσημα που έχουν σημειώσει την πορεία μας. Όταν ξεκίνησα εγώ πριν από 15 χρόνια, δεν ήταν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ο αθλητισμός. Παρ' όλα αυτά όμως προχωρήσαμε για να ε, ιδρύσουμε, για να χαιρετήσουμε το Ευρωπαϊκό Έτος της Εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού. Το χρηματοδοτήσαμε αφού είχαμε την αρμοδιότητα για την εκπαίδευση, έστω και αν δεν είχαμε αρμοδιότητες για τον ε, αθλητισμό προχωρήσαμε με το ευρωπαϊκό αυτό έτος και βήμα το βήμα μπορέσαμε να γεννήσουμε το αίσθημα ότι ναι, η Ευρώπη μπορεί να κάνει κάτι για τον αθλητισμό. Και με την πρόεδρό σας, την Doris Πακ, συνεργαστήκαμε στενά και μόνο έτσι μπορούσαμε να καταφέρουμε αυτή την πρόοδο και χάρη στην ε, ε, Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε την αρμοδιότητα και την αλλαγή των κανόνων. Αλλά πάντα βέβαια αναπολώ τα πρώτα αυτά χρόνια, τα πρώτα αυτά βήματα όπου κάποιοι προσπαθούσαν να μας αφήσουν εκτός του χώρου του αθλητισμού σε μια πρώτη συνάντηση με τους υπουργούς αθλητισμού δεν υπήρχε καν θέση για να καθίσει πρόεδρος της Επιτροπής και κάθισε, πήγα εγώ και πήρα μια καρέκλα και την έβαλα στη μέση των υπουργών του αθλητισμού και έτσι είχα ως επίτροπος ε, θέση να καθίσω στο τραπέζι των συζητήσεων. Και για τον πολιτισμό επίσης, με τη Helga Trüppel συνεργαστήκαμε για το Erasmus Mundus με τον κύριο Τάκουλα για την αδελφοποίηση πόλεων. Το Erasmus Mundus έχει αναπτυχθεί και μπόρεσα να δω και στο παιδί μου πρακτικά πώς λειτουργεί το Erasmus Mundus, 22 ετών και μπόρεσε πέρυσι να ε, εξασφαλίσει μια ανταλλαγή χάρη στο Erasmus Mundus ε, μεταξύ Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και Αμερικανικού και έτσι είδα ότι λειτουργεί το σύστημα αυτό και έτσι με χαρά διαπίστωσα ότι ένα βρέφος το οποίο ε, φέραμε στον κόσμο μεγάλωσε και λειτουργεί. Δεν μπορώ να σας πω πόσο σημαντικό είναι το Erasmus Mundus, όπως άλλωστε και η αδελφοποίηση των πόλεων που έχει και αυτή περάσει τη δοκιμασία του χρόνου. Και επίσης το δεύτερη μου θετία, κοινωνία των πληροφοριών και, των, και μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκεί απασχολη, μας απασχόλησε ιδιαίτερα η νομοθεσία, η νομοθέτηση. Είχαμε την οδηγία για τις ε, υπηρεσίες μέσω μαζικής ενημέρωσης, που αποτελεί ακόμη τη βάση της ε, τηλεόρασής μας και της ανάπτυξης του διαδικτύου, το Media Mundus και ένα πολύ δημοφιλές πρόγραμμα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιτεύχθη μια συμφωνία μεταξύ των χωρών που αποτέλεσε τη βάση της αναγνώρισης της ε, πολυπολιτισμικότητας όσον αφορά τις ε, κρατικές ε, επιδοτήσεις. Και σήμερα παραμένει η βασική αναφορά για τον κινηματογράφο, έστω με κάποιες αλλαγές. Ε, επίσης για το θέμα της δημοσιογραφίας ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και τέλος, την τρίτη μου θητεία ε, για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, το Ευρωπαϊκό Έτος για τον Εθελοντισμό, το Ευρωπαϊκό Έτος για τους ε, Πολίτες, το οποίο έχουν όλοι ακόμα κατά νου, γιατί το διευρύναμε από το 2013 στο πρώτο κομμάτι του 14 και συνέχισα να εργάζομαι για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας, πρόγραμμα το οποίο το μέλλον έχει εξασφαλιστεί και φροντίσαμε για την ε, τελική έγκριση στο Συμβούλιο, την οποία αναμένουμε και στη συνέχεια θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Ωραία λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει γερά θεμέλια, ούτως ώστε η μελλοντική γενεά να μπορεί να, να συνεχίσει την οικοδόμηση του κοινού μας οίκου έχουμε προάγει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα κοινό επίτευγμα και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Δεν ήταν το ένα θεσμικό όργανο το οποίο έκανε το ένα πράγμα και το άλλο κάτι διαφορετικό, αλλά πραγματικά ήταν ένα κοινό εγχείρημα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, προηγούμενους και τους ε, παρόντες ε, βουλευτές οι οποίοι συνεργάστηκαν για όλα αυτά τόσο στα επίπεδο της Επιτροπής όσο και στο Κοινοβούλιο γιατί πραγματικά το αποτέλεσμα το κερδίσαμε την Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ρέντινγκ. Πραγματικά αυτή ήταν μια πολύ καλή επισκόπηση ε, και πραγματικά όλοι λίγο πολύ συμμετείχαμε σε αυτό το εγχείρημα, σε ορισμένες δράσεις περισσότερο, σε άλλες ίσως όχι, αλλά ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, πού μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία στο μέλλον, το, το επόμενο έτος. Ωστόσο, είχαμε πολλές ε, δυνατότητες να συναντήσουμε τους νέους και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε εκεί όπου μπορούσαμε και πραγματικά είχαμε αποτελέσματα, μπορέσαμε να πετύχουμε ορισμένα αποτελέσματα, δεν στοχίσαμε σε, κάπα, σε κάποια άλλα, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια. Σαν Διάγο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ Ντόρις Ευχαριστούμε πολύ κυρία Αντιπρόεδρε που παρευρίσκεστε εδώ. Νομίζω ότι είναι πράγματι πολύ σημαντική αυτή η εκστρατεία που κάνετε σε διάφορους χώρους για να προάγετε το έργο της Επιτροπής και ιδιαίτερα την συμμετοχή στις προσεχείς ευρωεκλογέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που θα πάτε σύντομα στη Βαρκελόνη που είναι η δική μου πόλη γιατί νομίζω ότι εκεί είναι ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία σας και πιστεύω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξουν κάποιες εκλογές όπου θα γίνει λόγος για ευρωπαϊκά θέματα. Στην Καταλωνία υπάρχει, ε, γίνεται συζήτηση για μια ενδεχόμενη αυτονόμηση της ε, Καταλωνίας και ίσως αυτό το θέμα θα μονοπολίσει τις ευρωεκλογές και στο μέτρο αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό με μια προσωπικότητα όπω εσύ, η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορέσει να μεταβεί εκεί για να μιλήσει για τα σημαντικά ευρωπαϊκά θέματα και να τονίσει τη σημασία που έχουν γιατί αυτές οι εκλογές δεν θα πρέπει να εξυπηρετήσουν άλλους ε, στόχους, αλλά θα πρέπει να προαγάγουν τα ευρωπαϊκά θέματα τα οποία αφορούν ε, τους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί εγώ είμαι νέος βουλευτής αυτή τη θεατία και δεν είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σας ως ε, επίτροπος στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής, αλλά πραγματικά προωθήθηκαν σημαντικά πολλά θέματα στην Επιτροπή, ιδιαίτερα όσον αφορά τον αθλητισμό όπου εγώ έχω εθικευτεί κάπως περισσότερο και που είχα την τιμή να είμαι εισηγητής της πρώτης έκθεσης για τον αθλητισμό που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπως ε, είπατε εσείς ε, είστε... Ε, ναι, εντάξει, με διορθώνει η πρόεδρος ότι πρώτη και δεύτερη έκθεση, όχι την πρώτη. Ε, και ήταν, είναι ένα θέμα πραγματικά κεντρικής σημασίας σε αυτή την Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω που υπήρξατε πρωτοπόρος μαζί με την πρόεδρό μας, την κυρία Πακ, σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, Σαντιάγο, αλλά την πρώτη έκθεση για τον αθλητισμό την έκανα εγώ και στην έκθεση αυτή ε, ζήτησα πράγματα τα οποία συνέχεια εκπληρώθηκαν με τη Λισαβόνα. Εγώ τότε ήθελα ήδη να υπάρξει το έτος για τον αθλητισμό και όπως είπε η κυρία Ρέντινγκ κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να γίνει αλλά θα έπρεπε να το περιγράψουμε με πολλά λόγια για παράδειγμα το έτος της εκπαίδευση της αγωγής μέσω του αθλητισμού κλπ. κλπ. Αλλά τελικά το πετύχαμε. Αλλά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 Νομίζω ότι αυτός μπορεί να είναι ο, η, επιτυχία των εκλογών, ότι δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσουμε αυτά τα επιχειρήματα που προσπαθούν να ε, καταπολεμήσουν την εμβάθυνση στην Ευρώπη. Και αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Επίτροπε. Στο θέμα της προσέγγισης των πολιτών και στη δουλειά που γίνεται με τους πολίτες. Έχουμε και ε, στα προγράμματα για τον αθλητισμό, στα προγράμματα για την νεολαία. Έχουμε να κάνουμε 500 εκατομμύρια αποδέκτες πολίτες. Άρα λοιπόν πώς θα τους ε, μιλήσουμε, πώς θα στραφούμε σε αυτούς, εσείς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και εμείς στο δικό μας το επίπεδο επικοινωνίας και στις κοινέ μας ευθύνες μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βέβαια και με συμμετοχή των αρμόδιων για την επικοινωνιακή πολιτική ε, υπουργών, πώς μπορούμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα της Ευρώπης. Γιατί έχουμε προβλήματα σε αυτό το επίπεδο. Λιθουανία, ε, Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία. Ε, έχουμε πάρα πολύ μικρή ε, επαφή με τον κόσμο. Πώς μπορείτε λοιπόν να πείσετε και το Συμβούλιο ότι πρέπει να γίνεται καλύτερη επικοινωνία, επικοινωνιακή πολιτική και σε επίπεδο κυβερνήσεων. Αυτό πρέπει να το περάσουμε το μήνυμα. Και πρέπει να πείσουμε πόσο πολύτιμος αυρός είναι η Ευρώπη, πόσο σημαντικές οι, σημαντικά τα επιτεύγματα που μας έχει φέρει και πρέπει πιστεύω να ασκήσουμε και πίεση ακόμη προς τις κυβερνήσεις. Μπορείτε να το κάνετε εσείς αυτό κύριε Επίτροπε. Kiitoksia ja Kiitos. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την εξαίρετη παρουσίασή της και πραγματικά σκεφτόμουν ότι όταν βλέπουμε την πολιτική της Επιτροπής και κάνουμε τις σχετικές σκέψεις, νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε ούτως ώστε οι πληροφορίες να είναι ξεκάθαρες, να υπάρχουν λιγότερες πληροφορίες αλλά να είναι πιο αποτελεσματικές. Ε, και ο τρόπος που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενδέχεται αυτές τις πληροφορίες, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά όσο μιλούσατε, εγώ σκεφτόμουν ότι Έχουμε ορισμένε επιτυχίες, το Εράσμους, αλφαποίηση των πόλεων, τα αθλητικά προγράμματα, η Ευρώπη των πολιτών, ε, δημιουργώντας την Ευρώπη, πολλά προγράμματα τα οποία έχουν δώσει προσθέμενη αξία στην Ευρώπη και στην νεολαία. Και έτσι λοιπόν θα μπορούσα να πω ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να τονίσουμε αυτές τις ε, πολιτικές γιατί αναφερθήκατε στο θέμα των ευρωεκλογών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ θα ενδιαφέρονται ενδεχομένω για αποτυχίες, για μια αρνητική προεκλογική εκστρατεία. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε τις, τα πολλά επιτεύγματα, τις επιτυχίες της ε, Ευρώπης γιατί ορισμένες επιτυχίες θεωρούνται σαν αυτονόητες. Δεν τους προσδίδουμε αρκετή αξία, δεν τονίζουμε αρκετά όλα αυτά τα επιτεύγματα. Έχουμε εδώ κάποιους επισκέπτες από την Αυστραλία και αυτό δείχνει μία άλλη διάσταση των επιτυχιών μας. Είχαμε αυτή τη ε, συζήτηση, μπορούσαν να γίνουν αυτές τις συζητήσεις στα αγγλικά, στα γαλλικά κλπ. Τώρα μπορεί να γίνει ακόμα και στα φιλανδικά. Και αυτό πραγματικά είναι ένα επίτευγμα, γιατί πρόκειται για μια δύσκολη γλώσσα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω των. Ε, ξεπερνώντα τα γλωσσικά ε, σύνορα, του γλωσσικού φραγμού. Και αυτό δείχνει ότι μπορούμε να είμαστε ενωμένοι μέσα στι διαφορέ μα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, καλησμέρα σας ε, κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ανταλλαγή απόψεων που θεωρώ ότι είναι αναγκαία ούτως ώστε να τονίσουμε ε, τα κρίσιμα, τα επίμαχα σημεία αλλά και τις επιτυχίες ε, στο πλαίσιο αυτής της θητείας. Και πραγματικά έχετε δίκιο που αναφερθήκατε στην σημασία της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Και εδώ θα έπρεπε να θέσουμε το ερώτημα κάτω από το πρίσμα των δημοσκοπήσεων που έγιναν πριν από τις ευρωεκλογέ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε σχέση με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε, που ασκούμε. Κατά πόσο δηλαδή αυτός ο πολιτικός ο λόγος, η πολιτική συζήτηση που έγινε για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια ήταν πράγματι κάτι το οποίο μπορέσαμε να προβάλλουμε στην κοινή γνώμη, να περάσουμε στους ε, πολίτες. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να εδρεωθεί στη συνείδηση των πολιτών. Και αυτό το λέω γιατί είχαμε πολύ καλή συνεργασία όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος για τον Εθελοντισμό και το οποίο πραγματικά πρόκειται για ένα εξαιρετικό εργαλείο προώθηση με τέτοιου είδους ε, πρωτοβουλίες. Αλλά διαρωτώ με κατά πόσο το 2011 ε, μπόρεσε πράγματι να δώσει μια όφηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ε, συλλόγους της Ενώσης των Εθελοντών. Ενδεχομένως ε, ίσως παρέμεινε στο επίπεδο της επικοινωνία και ενδεχομένως δεν είχε μια αυθεντική μια σχέση με το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Και αυτό το λέω γιατί συζητήσαμε προηγουμένως για τον πολιτή προπολογισμό και γνωρίζουμε το πρόγραμμα Ευρώπη για τον πολίτη ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ε, δεν ε, πρικοδοτήθηκε με περισσότερα κονδύλια, αλλά αντίθετα έγιναν εδώ περικοπές. Το 2014 βεβαίως ε, αυξήσαμε τα κονδύλια, αλλά μακροπρόθεσμα θα έχουμε λιγότερα κονδύλια. Και αυτό πραγματικά θα είναι δυσάρεστο, ιδιαίτερα για τους ε, πολίτες σε μια εποχή όπου ζητούμε μεγαλύτερη συμμετοχή του πολίτη, μια μεγαλύτερη συμμετοχή στον την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Και εδώ περικόπτονται τα κονδύλια για πρωτοβουλίες μέσω των οποίων οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να αισθανθούν κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να μας πείτε τη δική σας άποψη. Τι απαντήσεις μπορούμε να δώσουμε στους Ευρωπαίους ε, πολίτες στο πλαίσιο της ε, προεκλογικής εξαρτίας. Βεβαίως ερχόμαστε σε επαφή με τον πολίτη και ανεξάρτητα από τις ευρωεκλογέ και αυτό μας, ε, μας προκαλεί κάποια αμηχανία. Ο κύριος Μάκουλα. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, εγώ έχω πολλά ε, ερωτήματα, παρόλο που θα περισσότερο ένα. Θα ήθελα να ζητήσω τη γνώμη σας για το μέλλον, τόσο μέσο όσο και μακροπρόθεσμα. Θα ήθελα να ρωτήσω για το διαδίκτυο, το ίντερνετ. Αναφερθήκατε στο διαδίκτυο στην παρουσίασή σας και γι' αυτό λοιπόν βασιζόμενος και στην εμπειρία, βασιζόμενο μάλλον και στην εμπειρία που έχετε, ε, γιατί υπήρξατε και Επίτροπος Πολιτισμού και Εκπαίδευσης και υπό την ιδιότητά σας αυτή θα ήθελα να σας ζητήσω τη γνώμη σας για την εξέλιξη του διαδικτύου ε, τόσο βράχη πρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Ε, και με αυτό εννοώ την πολιτική ενημέρωσης αλλά και αυτό το οποίο κάνει η δική μας Επιτροπή για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. Γιατί θέτω αυτό το ερώτημα, γιατί το ίντερνετ μέχρι ε, είναι το εργαλείο το οποίο έφερε τις περισσότερες αλλαγές στη ζωή των πολιτών τα τελευταία χρόνια. Και εγώ έχω αυτή την αίσθηση, γιατί προέρχομαι από μια χώρα, τη Ρουμανία, όπου βεβαίως υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά όσον αφορά το διαδίκτυο έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι. Και ε, σε μία έκθεση Net Index η οποία βασίζεται σε δεδομένα η οποία μελετά, εξετάζει την ταχύτητα των δεδομένων η Ρουμανία βρίσκεται σε πολύ καλή ε, θέση. Πέντε ε, πόλεις της Ρουμανίας βρίσκονται μεταξύ των δέκα πρώτων πόλων όσον αφορά ταχύτητα πρόσβαση στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν υπάρχουν χώρες που είναι τεχνικά εξοπλισμένες ούτως ώστε να μπορούν να αντλούν αυτές τις πληροφορίες από το διαδίκτυο και με τον τρόπο αυτό βεβαίως μπορεί να λειτουργήσει η επικοινωνία. Γνωρίζουμε βεβαίως τους κινδύνους που συνεπάγεται κάτι τέτοιο, τις ε, πληροφορίες οι οποίες ε, διαδίδονται, εξαπλώνονται και οι οποίες δεν είναι πάντοτε θετικές. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για το ίντερνετ καθώς και για την εξέλιξη του ίντερνετ από πολιστική αλλά και από νομική πλευρά γιατί εσείς είστε αρμόδια γι' αυτό. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Τρίπελ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στα θέματα του προπολογισμού και τα κονδύλια τα οποία προβλέπονται για την ε, πολιτική επικοινωνιών. Γιατί κατά την άποψή μου είναι πολύ απογοητευτό όταν μιλούμε για πολιτικέ επικοινωνιών και τονίστε πόσο σημαντικέ είναι να έχουμε μια περικοπή τάξη του 90% σε σχέση με την αρχική πρόταση ε, τη Επιτροπή. Και όταν βλέπουμε το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες και εδώ έχουμε δει περικοπή της του 23% και βεβαίω αυτό είναι πάρα πολύ αντιπαραγωγικό σε σχέση με τους στόχους τους οποίους έχουμε διατυπώσει. Γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε τη δική σας εκτίμηση για την κατάσταση αυτή και τα, την κατανομή των κονδυλίων. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ζαν Μαρή Καβαντά είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ πραγματικά ε, με συνδέει μια φιλία με την, την ε, πρόεδρο, με την κυρία Βίβιαν Ρέντινγκ. Αγαπητή Βίβιαν, ερχόμαστε από χώρες που πραγματικά ταλανίστηκαν από την ιστορία και εγώ και εσείς και εσείς κυρία Πρόεδρε και άλλες χώρες πιο πρόσφατα. Όταν βλέπουμε τα θετικά πράγματα που έκανε η Ευρώπη για να υποστηρίξει τις χώρες μέλη στις δυσκολίε τους πρόκειται για σημαντικά ποσά έστω και αν είναι διασπαρμένα ε, και τοποθετούνται σε διάφορα επίπεδα. Νομίζω ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια να διασωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία και αν δεν είχε γίνει αυτό θα είχαν περιέλθει μια κρίση πολύ χειρότερη από την κρίση του 1929. Αλλά υπήρξε τεχνοκρατική σε κάποιες λεπτομέρειες, κάτι το οποίο αποθαρρύνει τους Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι η βοήθεια την οποία έδωσε η Ευρώπη προς τις χώρες μέλη δεν γίνεται κατανοητή από την κοινή γνώμη σαν ένα εργαλείο υποστήριξης της λειτουργίας της στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης ε, έμαθα πολλά κυρία Ρέντινγκ από τη δική σας χώρα από τον Πιέρ Βερμέρ, τον Γκαστοντών, τον Ζαν Κλοντ Juncker και ορισμένες άλλες σημαντικές ε, προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων συμπαλαμβάνεστε και εσείς, κυρία Ρέντινγκ. Ε, και πραγματικά ήταν ε, πολύ σημαντικό για αυτή τη γενεά δεν υπάρχει ούτε ένας... Ε, στη, στη, Γαλλία είναι μόνο ένας στους δύο πολίτες που προσέρχεται στις ε, κάλπες, γιατί δυστυχώς δεν είναι υποχρεωτικές ε, οι εκλογές. Άρα λοιπόν υπάρχει μια απομάκρυση μεταξύ του απολογισμού των επιτεγμάτων της Ευρώπης και της αντίληψης που έχει ο πολίτης ή της Ιδέα που έχει ο πολίτης για όλα αυτά. Δεν θα ήθελα να υποτιμήσω τις δικές σας προσπάθειες, κυρία Ρέντινγκ, προς την κατεύθυνση αυτή. Παρ' όλα αυτά δεν ε, βλέπουμε απτά τα αποτελέσματα σε σχέση με την αναγνώριση της κοινή ε, γνώμης όσον αφορά τα επιτεύγματα της Ευρώπης. Άρα λοιπόν ε, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη καμπή. Ακόμα και στη χώρα μου από την οποία προέρχομαι εκεί το βάρος των αντιευρωπαϊστών οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι δημοκράτες αλλά στην πραγματικότητα είναι υπέρμαχοι μιας βίαιης πολιτικής και περιμένουν πραγματικά να ανέλθουν στην εξουσία για να επιβληθούν και όχι να λειτουργήσουμε μέσω της δημοκρατικής πυθούς. Βεβαίως, τα ε, θεσμικά όργανα είναι παραχωμένα, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των επιτρόπων, δεν είναι αρκετά μεγάλο το κύρος ε, των οργάνων αυτών στο Συμβούλιο. Και πέρα από αυτά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτως ώστε να βρούμε σημαντικούς Ευρωπαίους ηθήνοντες οι οποίοι ε, είναι αρκετά θαραλέοι και δεν ε, υπεκφεύγουν χρησιμοποιώντας την Ευρώπη σαν ε, ασπίδα για τα δικά τους συμφέροντα. Γιατί πραγματικά αυτό θα ήταν μια αληθινή καταστροφή. Εδώ και δύο θητείες σας βλέπω να ασκείτε τα καθήκοντά σε δύο γειτονικούς τομείς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία είναι επιτυχία, ενώ αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουγγαρία είναι καταστροφικά. Αυτό είναι λάθος να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις. Πώς μπορούμε να καταφέρουμε ούτως ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να αποφύγει αυτό το, την ε, διάσταση της ε, βαρβαρότητας, αλλά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ε, προωθώντας τον πολιτισμό και τα πολιτισμικά αγαθά και όχι τις αξίες της βαρβαρότητας. Ευχαριστώ. Έχω μερικέ παρατήρησει να κάνω και εγώ από τη δική μου πλευρά. Να τι κάνω, λέει κυρία Πάκ. Θα ήθελα να χαιρετήσω καταρχήν το γεγονό ότι έχουμε το Europe Direct, όπου νομίζω ότι γίνεται πολύ καλή εργασία ε, είναι ουδέτερη πολιτικά, είναι πολύ χρήσιμη τα... και οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ καταρτισμένοι και πραγματικά είμαι ευγνώμων που στη δική μου πατρίδα, στο Ζαρμπρούκεν, αυτό το Europe Direct κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχω επίσης την άποψη ότι το εγχειρίδιο για τα δικαιώματα των πολιτών σίγουρα είναι χρήσιμο για μας και ίσως θα ήταν χρήσιμο αν μπορούσε να υπάρχει, να διατίθεται σε πολλές γλώσσες και ίσως θα ήταν χρήσιμο να ξέραμε από πού μπορούμε να το βρούμε. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα να πάει κανείς στην ε, Πολωνία ε, και οι Πολωνοί να μιλούν ε, αγγλικά. Ε, χρήσιμο είναι να υπάρχουν ε, τα χερίδια αυτά στη γλώσσα ε, της κάθε χώρας. Τρίτον, το Europe Around the Corner. Ε, μου φαίνεται μια καλή μεν ιδέα γιατί αυτό βοηθάει τους συναδέλφους να ξέρουν τι είναι αυτό το οποίο προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, αλλά και θα πρέπει πραγματικά αυτές οι συστάσεις να φτάνουν στους συναδέλφους. Ίσως θα ήταν καλό να μας δώσετε ένα κείμενο που να λέει πού μπορούμε ακριβώς να αντλήσουμε αυτές τις πληροφορίες, που βρίσκουν, που διατίθενται αυτές τις πληροφοριες που βρισκονται που διατιθενται αυτες τις πληροφοριες Και έχω και μία άλλη ερώτηση για τη νέα αφήγηση, το new narrative, για την οποία μιλήσατε. Αυτή ήταν η ιδέα του συναδέλφου κυρίου Λόκαγκατ, ανεξάρτητα από την Επιτροπή Πολιτισμού και η οποία συμπελήφθη στον προπολογισμό και από ο κύριος Μπαρόζο και ο Βασίλειο τελικά ε, ε, στο οποίο αντέδρασαν με χαρά. Αλλά σε αυτό, αυτό είναι κάτι μια έννοια στην οποία αναφέρονται οι φιλόσοφοι, οι καλλιτέχνες, την έννοια της νέας αφήγησης αλλά δεν θα βρείτε μεταξύ αυτών βουλευτές, θα βρείτε στον τον κύριο Λόκεγκαρτ ή την κυρία Πακ υπό την ιδιότητά τη ω Προέδρου αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε την ε, δυνατότητα αυτή η δεξαμενή σκέψη, η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει να δίνει σε περισσότερους συναδέλφους να έρθουν μαζί της σε επαφή. Η τελική συνδιάσκεψη θα γίνει στην, ε, την 1η Μαΐου στο Βερολίνο και δεν είμαι καθόλου σίγουρη αν έχει προσκληθεί κάποιος άλλος εκτός από τον κύριο Λόκγκαρτ και εμένα. Ε, και νομίζω ότι αυτό δεν είναι εξαιρετικά βοηθητικό. Εάν ε, λέτε ότι θέλουμε να συναντηθούμε με στοχαστές, ε, με διανοούμενους και καλλιτέχνες, τότε νομίζω ότι θα έπρεπε να δοθεί και στους συναδέλφους ευκαιρίες, η ευκαιρία να παρευρεθούν. Ε, την 1η Μαρτίου, όχι Μαΐου. Την 1η Μαρτίου λοιπόν στο Βερολίνο θα διοργανωθεί το τελικό συμπόσιο στο Βερολίνο. 1η Μαρτίου λοιπόν στο Βερολίνο και αν ενδιαφέρεστε θα φροντίσω να προσκληθείτε γιατί θεωρώ θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να παρασταθείτε. Και δύο άλλες παρατηρήσεις. Και εμάς μας λείβει το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της δικής σας ε, θητείας ε, χάθηκαν κάποια πράγματα στην αρχή, αλλά αυτό έχει πάρει πολύ καιρό από τότε. Στην αρχή, όταν ξεκινήσατε, η Επιτροπή είχε την, ε, κατέστρεψε την ε, Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών ε, Σπιτιών. Αυτό πραγματικά ήταν ένα πραξικόπημα και ακόμα υποφέρουμε από τις συνέπειες αυτού του πραξικόπηματος. Το άλλο είναι ότι το Euronet, το ραδιοφωνικό δίκτυο, μπορέσαμε να το διατηρήσουμε με πολλούς κόπους. Το έχουμε μεν, αλλά χωρίς το Κοινοβούλιο δεν ε, πρόκειται να υποστηριχθούν. Και το τρίτο στοιχείο είναι το εξής. Δεν ε, υπάρχει πλέον το diary, ε, το οποίο επιζητούν πάρα πολύ, γιατί και, και αυτό δεν υποστηρίχθηκε με κονδύλια από την Επιτροπή. Υπάρχουν πάρα πολλοί δάσκαλοι που έχουν απευθυνθεί σε μένα λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για το μάθημα, γιατί το καταργήσατε. Και το τελευταίο, ο Ροπρές, το οποίο έδωσε μας την ευκαιρία, το Europress, ε, να διαβάζουμε τι γράφει ε, στις 28, στα 28, στις 28 χώρες στον τύπο για ένα θέμα. Να μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι απόψεις του τύπου για ένα θέμα σε όλες τις χώρες μέλη, το Europress. Και αυτό δεν υποστηρίχθηκε με κονδύλια. Και θα πρέπει να το πω γιατί πραγματικά πάρα πολλοί απευθύνονται σε εμά λέγοντας γιατί καταργήσατε όλα αυτά. Και θα ήθελα να πω ότι μας θλίβει γιατί πολύ συχνά ε, τελικά προσπαθούν να ξαναφεύρουν τον τροχό χωρίς να θέλουν να συνεχίσουν τη λειτουργία κάποιων άλλων πραγμάτων που ήταν ιδιαίτερως ε, πετυχημένα, μόνο και μόνο για να επινοήσουν κάποια νέα. Και πραγματικά ως πρόεδρος αυτής της Επιτροπής αισθάνομαι υποχρεωμένη να αναφερθώ και σε αυτά τα θέματα γιατί πραγματικά ήταν πολλές προσπάθειες τις οποίες ε, χαιρετήσαμε αλλά υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα ε, τα οποία καταργήθηκαν και υποφέρουμε ακόμα από τη συνεπείς της εξαφάνισής τους. Και ε, τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Βίβια. Όχι, συνάδελφος κυρία Ντουμπρόβκα από το Um, uh, Δεν ξέρω αν ε, είναι στο χαρτοφυλάκιο της κυρίας ε, Ρέντινγκ για η δικαιοσύνη και η θαγένεια αλλά να ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με την Επιτροπή μας. Είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Δεν ξέρω, ίσως γνωρίζει λίγα παραπάνω η κυρία Ρέντινγκ. Έχω κάνει την ερώτηση αυτή. Ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα ε, μεταξύ των δύο συνομοθετών, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Το έχουμε λύσει αυτό, δεν υπάρχει πια πρόβλημα, έχει διεκπεριωθεί και καμία σχέση πλέον με την κυρία Ρέντινγκ. Στο μεταξύ δεν είναι αρμόδια για το πολιτισμό, είναι η κυρία Βασιλείου. Και έχει να κάνει κάτι με το δικό μας τριμερή διάλογο, ο οποίος τώρα τελειώνει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη. Όλα εντάξει είναι, μην ανησυχείτε. A lot of uh, Έγιναν πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όσο γίνεται ε, και ε, όσο τις σημείωσα. Ο διάλογος των πολιτών στη Βαρκελόνη. Βεβαίω και θα είναι δύσκολος, αλλά θα είναι διαφορετικός από τους προηγουμένους. Έχω ζήσει πολλούς δύσκολους διαλόγους και ήταν όλοι διαφορετικοί μεταξύ τους. Συστηματικά Κάθε φορά που πηγαίνω στο Νότο, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, Ισπανία ε, και ε, συζητούσαμε εκατοντάδες νέων. Ο διάλογος με τους πολίτες είναι ερωτήσεις, απαντήσεις, καμία σχέση με ομιλίες ενώπιος ενωπίο και πρέπει να σας πω ότι πολλοί διάλογοι ήταν πάρα πολύ σκληροί και στη Σόφια θυμάμαι ένα, όπου ο κόσμος περίμενε τέσσερις ώρες την ουρά για να μπει και τελικά ε, είχαν για πρώτη φορά πολιτικούς που μπορούσαν να τους μιλήσουν απευθείας, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε μένα. Και άρχισαν να φωνάζουν. Όχι σε μένα, αλλά ε, γιατί απλούστατα δεν είχαν άλλη ευκαιρία να απευθυνθούν ε, άμεσα στη Βουλγαρία σε πολιτικούς πλέον. Και μετά από το διάλογο αυτό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εθέσπισε αυτό το διάλογο παντού στη χώρα. Και υπάρχει πίεση πλέον πολύ μεγάλη σε δύσκολες περιφέρειες για τους ε, Δικού του πολιτικούς και σου λένε γιατί θα πρέπει να έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσει και να μας απαντήσει. Ορίστε, καθίστε κι εσείς να μας ακούσετε και να μας δίνετε εσείς τις απαντήσεις. Αυτοί οι διάλογοι λοιπόν ε, πολλαπλασιάστηκαν και ήταν και πολύ διδακτικοί για μένα την ίδια. Ε, να σας δώσω δύο διδάγματα που αποκόμισα. Παντού Βέβαια κάθε διάλογος είπαμε ενδιαφέρει. Φανταστείτε στο Λονδίνο αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η ελεύθερη κυκλοφορία κυρίως. Στην Ελλάδα είχε να κάνει περισσότερο με το υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ. Η χώρα αυτή θα συνεχίσει να ζει. Πώς θα μας βοηθήσετε. Στη Γερμανία ε, ήταν πολύ ε, λόγος για τα δικαιώματα των πολιτών με κάθε μορφή. Ε, δεν ήταν ένας ο διάλογος δηλαδή. Άλλοι μου είπαν μην ανακατεύεται πάρα πολύ η Ευρώπη. Μάλλον το περίμενα γιατί το λέει ο τύπος. Μόνο ο τύπος το λέει όμως, οι πολίτες όχι. Οι πολίτες δεν θεωρούσαν ότι αυτό είναι θέμα. Το αντίθετο. Επανειλημμένα χρειάστηκε να εξηγήσω σε πολίτες γιατί δεν μπορούσαν να κάνω κάτι και με ρωτούσαν. Γιατί. Και οι απαντήσεις ήταν ότι είναι στη συνθήκη. Και η απάντηση των πολιτών ήταν να την αλλάξει τη συνθήκη για να μου λύσει το πρόβλημα. Γενικά λοιπόν οι πολίτες θέλουν να λύνονται τα προβλήματά τους και δεν τους ενδιαφέρουν οι θεσμικές μας κατασκευές. Θέλουν έναν που να τον εμπιστεύονται και αυτός να μπορεί να λύνει τα προβλήματά τους. Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία ή το πρώτο δίδαγμα. Και ένα δεύτερο για τις ευρωεκλογέ. Με την εξαίρεση του Λουξεμβούργου, που είναι άλλη ιστορία του Λουξεμβούργου, κόσμος δεν έχει ιδέα για τους ευρωβουλευτές, δεν τους γνωρίζουν. Δεν ξέρουν ούτε τι κάνει το κοινοβούλιο, ούτε τι εξουσίες έχει το κοινοβούλιο. Σε κάθε διάλογο, τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά πρέπει να αφιερώνω για να εξηγώ ποιες είναι οι μεγάλες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συναποφασίζει, συνομοθετεί οι νόμου που στη συνέχεια εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Ο κόσμος δεν τα γνωρίζει αυτά απλούστατα. Και γιατί σας το λέω διότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό θα έρθετε αντιμέτωποι στην προεκλογική εκστρατεία με πολλούς που δεν έχουν ιδέα. Και ένα από του λόγους που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν στι ευρωεκλογέ οι πολίτες είναι διότι δεν ξέρουν για ποιο λόγο να πάνε, τι τους αφορά αυτό και τι ε, εξουσία έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο έχω πάρει από παντού. Με εξαίρεση, επαναλαμβάνω, το Λουξεμβούργο. Οι Λουξεμβούργοι είναι οι μόνοι που γνωρίζουν τι εστί Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γιατί ο τύπος ε, στο Λουξεμβούργο συνεχώς αναφέρει ε, τι κάνουν στις Βρυξέλλες οι Ευρωβουλευτές και στο Στρασβούργο. Λοιπόν, ευρωσκεπτικισμός. Νομίζω ήδη το αναφέραμε και αυτό. Έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το εξής. Και οφείλεται στο γεγονός ότι ε, οι, πολιτικές, οι πολιτικοί στα κράτη-μέλη δεν εξηγούν ποτέ τι γίνεται στην Ευρώπη. Προσπαθήστε να κάνετε λίγο ζάπινγκ στην τηλεόραση μετά από μια συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες σε διάφορα κανάλια ειδήσει, τι λέγουν και τι αναφέρουν και πώς μεταφέρουν για το τι έκανε ο υπουργό ή ο Πρωθυπουργό του στις Βρυξέλλες. Και μετά τι εξηγεί ότι έκανε ο υπουργό ή ο Πρωθυπουργό. Κανονικά έχει ως εξή. Πήγα στις Βρυξέλλες και κέρδισα. Του τάπα. Δηλαδή εγώ κέρδισα και άλλοι χάσανε. Και ευτυχώ ήταν αρκετά ισχυροί οι υπουργοί τη εκάστοτε χώρα για να παραγκονίσουν όλου του άλλου. Δεν υπάρχουν υπουργοί και πρωθυπουργοί που να λέγουν Ξέρετε ποια είναι τα προβλήματα, ξέρετε γιατί θέματα συζητήσαμε. Ευτυχώ βρήκα πολλού συμμάχου από την τάδε τη δίνα χώρα και μαζί καταφέραμε να περάσουμε την εξή ιδέα. Ποτέ δεν θα ακούσετε τέτοιο πράγμα από υπουργό σε καμία γλώσσα στην Ευρώπη. Και αυτό είναι πρόβλημα. Πώς ξαφνικά μπορεί η Ευρώπη να γίνει σημαντική στα μάτια των πολιτών, δημιουργική, να κάνει κάτι για τους πολίτες, όταν στο τέλος η Ευρώπη την οποία εξηγούν οι υπουργοί στους οποίους οι πολίτες έχουν εμπιστοσύνη είναι μια Ευρώπη στην οποία θα πρέπει να μπει ένα φρένο και το έβαλαν οι ίδιοι πηγαίνοντας στο Υπουργικό Συμβούλιο και επιβάλλοντας τις απόψεις τους. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Ορισμένοι με ρώτησαν πώς συνεργαζόμαστε τα διάφορα θεσμικά όργανα. Πρέπει να σας πω ότι η συνεργασία μας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ως εξής. Πολύ συχνά στα κράτη-μέλη έχουμε τους λεγόμενους οίκους της Ευρώπης, ε, με λερό που είναι τα γραφεία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, στην ίδια στέγη και σε διοργανώνουν ε, δραστηριότητες και πηγαίνουν καλά τα πράγματα τις περισσότερες φορές. Εκεί που δεν πηγαίνουν τόσο καλά είναι στη συνεργασία με τις κυβερνήσεις. Έχουμε ε, συνεργασίες για διαχείριση διαφόρων προγραμμάτων και θεμάτων και στα χαρτιά έχουμε και κοινά ε, σχέδια επικοινωνίας. Αν ενδιαφέρεστε, έχω φέρει να σας πω ποια είναι τα προγράμματα αυτά και τι κάνουμε. Σε δύο κράτη-μέλη Δύο από 28 κράτη-μέλη, το Βέλγιο και η Αυστρία, συγχρηματοδοτούν αυτά τα προγράμματα. Και δύο ή τρία κράτη έχουν μια συμβολική συνεισφορά, αλλά όχι ουσιαστική για να λειτουργούν όλα αυτά. Δεν θέλω να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, αλλά έχουμε πραγματικό πρόβλημα ε, με τη συνεργασία των κρατών μελών όχι τη θεωρητική, την ουσιαστική και την πρακτική. Για να ε, μπορέσουν αυτές οι σχέσεις ε, εταιρικέ να λειτουργήσουν. Δεν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη ε, για την κατάσταση αυτή, αλλά έτσι έχει. Να βρούμε μια απλή γλώσσα για τους πολίτες. Α, τα θεσμικά όργανα υπάρχουν και οι θεσμοί γενικά. Το Europe Direct κάθε χρόνο δέχεται ένα εκατομμύριο ερωτήσεις αυτής επεξεργάζεται και δίνει κάποιες απαντήσεις στους πολίτες σε απλή γλώσσα. Έχουμε 500 γραφεία ε, για το σκοπό αυτό με καταρτισμένο προσωπικό για την προεκλογική εκστρατεία ε, και ξέρουν να απαντήσουν και στα δύσκολα, στα καθόδια ερωτήματα και ξέρουν πού να αποτανθούν για να πάρουν απάντηση. Θα ενημερώσουμε και το Κοινοβούλιο για το νέο πρόγραμμα Europe Around the Corner πριν τις εκλογές. Η Ευρώπη δίπλα σας, σε όλες τις γλώσσες δηλαδή, για να μπορούν ε, και ένα εγχειρίδιο θα μοιραστεί. Δεν είναι πολιτικό, είναι πάρα πολύ απλό για τα δικαιώματα ε, που παρέχει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολύ σαφή γλώσσα και απλή. Τουλάχιστον αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε και αυτό προσπαθούμε. Οι αρνητικέ εκστρατείε των μέσων ενημέρωση, όσοι γνωρίζουν ε, περί δημοσιογραφίε, ξέρουν ότι οι καλέ ειδήσει δεν είναι ειδήσει. Άρα τα κακά νέα πουλάνε. Αν εσεί ως βουλευτές παράγετε κακές ειδήσει, είστε βέβαιοι ότι θα μπείτε στο δελτίο ειδήσεων. Παράδειγμα, την περασμένη Δευτέρα, τώρα, προχτές, ήμουν σε ένα διάλογο πολιτών στο Λονδίνο. Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό, ότι ήταν δύσκολη η κατάσταση και ε, πολύ μεγάλες δυσχέρεις. Ε, την ώρα που ήμουν εγώ στο διάλογο των πολιτών, μου κλείψαν τις αποσκευές μου. Τι έγραψε ο τύπος για το διάλογο για το δύσκολο διάλογο, για τους αγώνες που δίνουμε για την ελεύθερη κυκλοφορία. Όχι. Όλοι έγραφαν ότι μου κλέψαν τις αποσκευές. Είχες και τα σκουλαρίκια σου μέσα και διάφορα κοσμήματα, ναι. Ναι. Ε, τι να κάνει κανείς, ε, έτσι έχει ζωή, έτσι έχουν τα μέσα ενημέρωση. So, Uh, the, uh, the, the worry Η ανησυχία ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν τι σημαίνει η ηθαγένεια είναι πραγματική ανησυχία. Το ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι τα τέσσερα πέμπτα των πολιτών μας, κατά μέσον όρο, γιατί υπάρχουν αποκλήσεις από κράτος σε κράτος, γνωρίζουν κατά μέσον όρων λοιπόν ότι είναι ε, Ευρωπαίοι και αισθάνονται Ευρωπαίοι, αλλά μόνο ένα τρίτο των πολιτών γνωρίζει τι σημαίνει αυτό. Θα ήθελα να έχουν περισσότερη πληροφόρηση και συνήθως δεν ξέρουν και πού να στραφούν για την πληροφόρηση. Ακόμα και αν τους βάλει κανείς το χέρι, δηλαδή το φυλάδιο για όλες τις δυνατότητες ενημέρωσης που διατίθενται, δεν τις αξιοποιούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί θα έχει χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα η εκλογική εκστρατεία γιατί θα δείξει στους πολίτες πώς μπορούν, από πού μπορούν να αναστήσουν τις πληροφορίες. Ε, τα διάφορα ευρωπαϊκά έτη του εθελοντισμού, της ηθαγένειας κτλ. που οργανώνουμε έχουν σημασία για να περάσει το συγκεκριμένο μήνυμα αλλά ταυτόχρονα και με όλες τις ενημερωτικές δραστηριότητες και τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε στη συζήτηση και με όλα αυτά που κάνουμε πάλι είναι πολύ περιορισμένο το ποσοστό των πολιτών που ε, δείχνουν ενδιαφέρον και ακούνε τι έχουμε να τους πούμε. Και βεβαίως μπορούμε με το ίντερνετ να ενισχύσουμε την ενημέρωση. Σε έναν διάλογο πολιτών έχουμε περίπου 500 πολίτες μέσα σε μια αίθουσα συζήτησης, αλλά αρκετές χιλιάδες συνδεδεμένους μέσω του διαδικτύου που παρακολουθούν ζωντανή τη συζήτηση από το streaming και άλλους που επικοινωνούν μέσω του Facebook και του Twitter. Άρα μπορούμε χάρη στα μέσα αυτά να περάσουμε καλύτερα το αποτέλεσμα. Και έχοντας αναπτύξει και διαδικτυακό διάλογο, chat, με τον οποίο βέβαια μπορεί κανείς να προσεγγίσει πολύ περισσότερο κόσμο από ότι μέσα σε μια αίθουσα συνεδρίασης. Ε, ξέρω ότι μπορεί αυτό το νέο μέσον, το, ο κόσμος αυτός ο νέος του ίντερνετ να ενισχύσει την επικοινωνία. Αλλά παρόλα κρύβει και προβλήματα. Η Επιτροπή σας, αν δεν απατώμε, είναι εκείνη η οποία έχει συζητήσει πολύ το θέμα του ασφαλέστερου διαδικτύου, διότι υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι ε, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να επιβουλευθούν την ασφάλεια των παιδιών μας. Και πρέπει το διαδίκτυο να το προωθήσουμε, ενημερώνοντας όμως και τους γονείς για το τι είδους κινδύνους αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους από το διαδίκτυο. Επίσης, Έχουμε την μεταρρύθμιση των, της νομοθεσίας για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που έχει συμβάλει πολύ το Κοινοβούλιο γιατί ψήφισε με συντριπτικές πλειοψηφίες νέους κανόνες πιο καλά προσαρμοσμένους στο νέο διαδικτυακό κόσμο. Το Συμβούλιο όμως των Υπουργών δεν έχει ακόμη ε, καταλήξει, δεν έχει μπορέσει να λάβει τις πολιτικές αποφάσεις που θα έπρεπε να λαμβάνει. Και εάν δεν συνεργάζονται τα τρία θεσμικά όργανα, προβλήματα θα έχουμε. Έχουμε πολύ συχνά πολύ καλή συνεργασία μεταξύ Επιτροπή και, και Κοινοβουλίου, αλλά το Συμβούλιο πολύ συχνά είναι εκείνο το οποίο προξένει τα προβλήματα και δεν μπορούμε να ε, κλείσουμε κάποια θέματα. Επίσης, λυπούμε που δεν έχουμε υψηλότερο προϋπολογισμό. αυτά τα οποία εγώ έχω υποβάλει σαν προτάσεις, τα αποφάσισαν διαφορετικά τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αποφασίστηκαν περικοπές και με αυτές τις περικοπές θα πρέπει να πορευτούμε. Μείον 15% για το πρόγραμμα για, τους, για την υπηκότητα, επικοινωνιακή πολιτική μείον 12%, ε, επίσης στην επικοινωνία μείον 9%, για τους πολίτες, Ευρώπη για τους πολίτες μείον 3%. Ε, όλα αυτά σημαίνουν περικοπές σημαντικές και πρέπει να, τις, ε, να προσαρμόσουμε τα προγράμματά μας με βάση αυτές τις περικοπές. Δεν μπορούμε να καταβάλουμε τα ποσά που θα θέλαμε. Δεν μπορούμε να καλύψουμε δηλαδή όλες μας ανάγκες και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε περικοπές σε ορισμένες περιπτώσεις ε, κατακόρυφα, δεν μπορούμε να κόψουμε ένα μικρό κομματάκι από κάθε πρόγραμμα, γιατί τότε θα τα εξοδερώναμε όλα, για να μπορέσουν να επιβιώσουν κάποια προγράμματα, χρειάστηκε να κάνουμε κατακόρυφες περικοπές σε κάποια άλλα. Για τα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματά σας για το Europe Direct απήντησα για τα δικαιώματα πίντησα, για το Europe Round the Corner. Θα είναι πληροφορία διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Θα σας ενημερώσω και γραπτός, ώστε να έχετε και τα links στους συνδέσμους και να τους ε, δώσετε στους συναδέλφους σας βουλευτές. A new narrative, νέα τοποθέτηση, νέα ορολογία, αφήγη. νέο αφήγημα ε, δεν έχει σχέση τόσο πολύ με τους βουλευτές όσο με την επικοινωνία με επιστήμονες, φιλοσόφους, καλλιτέχνες ώστε να διατυπώσουν εκείνοι τις προτάσεις τους. Αυτά είναι βασική ιδέα. Όταν όμως ετοιμάσουν τις προτάσεις τους και αυτοί θα πρέπει οι προτάσεις αυτές να δημοσιοποιηθούν. Ωστόσο πρόκειται για μια ε, συμβολή αυτή τη ομάδα των πολιτών, τη κατηγορία πολιτών που συνήθως δεν ρωτάμε τη γνώμη του. Και με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό δέχθηκαν να συμμετάσχουν. Χαίρομαι που προχώρησε αυτή η υπόθεση και περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τα πορίσματα των εργασιών τους για την 1η Μαρτίου, τα οποία θα αξιοποιήσουμε περαιτέρω. Έχουμε ήδη πολλές φορές μιλήσει για το Euronaut. Έχει διαφυλαχθεί και αυτό είναι καλό, αλλά η τροπολογία μόνο ένα έτος ε, λειτουργίας του καλύπτει, γιατί έγιναν σοβαρές περικοπές και άρα θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα ένα έτος. Οπότε θα πρέπει να δούμε με λιγότερα χρήματα πώς, πώς θα μπορέσουμε να α, κάνουμε να λειτουργήσουν συστήματα που έχουν πολλά χρήματα. Έχουν επενδυθεί στο Euronet τα χρήματα τα οποία μας έχουν διτεθεί για να μπορέσουν να λειτουργήσει. Επίσης ε, θα ήθελα να πω ότι η συνάδελφος Μίμικα ο... για το χρονοδιάγραμμα ο συνάδελφος ε, έχει ε, την αρμοδιότητα αυτή για το σχολικό έτος επίσης. Το Press Europa έχουμε πολλές φορές συζητήσει ξεκίνησε το 2008. Για ένα έτος έχει αναθεωρηθεί τέσσερις φορές το μέγιστο επιτρεπόμενο. Εξέπνευσε δε στις 22 Δεκεμβρίου του 2013. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε όχι αυτό αλλά κάποιο αντίστοιχο έργο. Εάν κάναμε μια προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος, μια νέα διαδικασία με ανοιχτέ υποψηφιότητε δηλαδή, λόγω έλλειψης κονδυλίων αποφάσισαμε να μην ξεκινήσουμε νέο έργο όμω. Γιατί δυσκολευόμαστε να διατηρήσουμε εν ζωή τα εν εξελίξει έργα. Αλλά η χρηματοδότησή μας και πάντοτε επέμενε σε αυτό το κοινοβούλιο, η χρηματοδότησή μας δεν έχει έναν χαρακτήρα ατέρμονο χρηματοδότησή μας έχει σαν ε, στόχο να δώσει το ε, ε, ένα κτίριο λάξιμο, να δώσει την όθηση για να ξεκινήσει ένα έργο, το οποίο μετά θα αυτοχρηματοδοτείται. Το έχουμε κάνει ήδη, έχουν ξεκινήσει ιδέες και μπορούν να συνεχίσουν εφόσον είναι καλά project, καλά έργα να απογειωθούν και να συνεχίσουν να λειτουργούν για κάποια χρόνια μόνο τους. Αυτά εν ολίγης, όσα είχα να σας πω. Η σημαντική σας επιτροπή και ο Ζωμανή Καβαντά το είπε πολύ σωστά πριν. Η Ευρώπη όχι μόνο της οικονομίας και του ευρώ, του χρήματος, θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, αλλά θα είναι και η Ευρώπη των ιδεών, των αξιών, των πολιτών. Η Ευρώπη αυτή που μπορεί η Επιτροπή σας και στο νέο Κοινοβούλιο να προβάλλει με στεναρό τρόπο, να είναι μια ισχυρή Επιτροπή και να αναπτύξει αυτό ακριβώς που περιμένουμε. Και αυτό είναι η αγορά, ε, όχι η αγορά, αλλά οι άνθρωποι. Ευχαριστώ. Η κυρία Τρίπελ έχει μια ερώτηση. Ναι, μια συμπληρωματική ερώτηση, κυρία Επιτροπέ, γιατί είπατε ότι συνήθως οι υπουργοί γυρνάνε στις πατρίδες τους για να ισχυριστούν ότι έχουν κερδίσει τον αγώνα στις Βρυξέλλες. Δεν έχετε σκεφτεί να βρείτε μία λύση εσείς από την Επιτροπή και κάποιοι πιο υπεύθυνοι από το Συμβούλιο να, κάνετε αυτή την, ε, να αναπτύσσετε αυτή την επικοινωνιακή πολιτική ώστε να δίνετε τη σωστή ενημέρωση. Να έχετε μια κοινή στρατηγική για την επικοινωνία. Κοιτάξτε, πολλοί από τους επιτρόπους θεωρούνται πολύ αξιόπιστοι στις πατρίδες τους. Από τις αναλύσεις που έχουμε κάνει βλέπουμε ότι λίγοι είναι οι επίτροποι όμως που μπορούν να βγουν σε οποιαδήποτε χώρα και να θεωρηθούν αξιόπιστοι. Οι περισσότεροι όμως στη δική τους την πατρίδα είναι πιστευτοί και ως εκ τούτου αξιοποιούνται, αξιοποιούν το μέσον της τηλεόρασης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη χώρα τους για να απευθυνθούν στους πολίτες. Και κάθε μέρα επίσης δημοσιεύουμε έναν τόμο ολόκληρο με άρθρα που απευθύνονται στον τύπο με συνεντεύξεις επιτρόπων. Κυρίως προς τα κράτη-μέλη αλλά και εκτός αυτών. Αυτό είναι σημαντικό. Άρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το μέσο της τηλεόρασης. Μπορεί να πει ένας ε, επίτροπος όμως «Α, όχι, αυτά που είπε ο Υπουργός είναι χαζομάρες και δεν ήταν έτσι». Όχι, όχι, δεν ήταν αυτή η ερώτησή μου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, συγκρούσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει τρόπος να συνδυάσετε το μήνυμα που απευθύνεται, να παρουσιάσετε συνδυασμένο το μήνυμα μαζί με τους υπουργούς και να δείξετε ότι υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ του εθνικού και του ευρωπαϊκού επίπεδου. Επειδή αναφερθήκατε σε αυτή τη ε, διαδικασία ε, επίρρυψης ευθυνών και κατηγοριών, δεν μπορείτε να το, την αντιμετωπίσετε με άλλο τρόπο. Πολύ ωραία η ιδέα σας και την επικροτώ. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι, ύστερα από 15 χρόνια εμπειρίας, με το Συμβούλιο των Υπουργών και τη συνεδριάσεις του, γιατί συνήθως παρακολουθώ ολόκληρη τη συνεδρία των Υπουργών, αλλά κάθε δέκα λεπτά οι υπουργοί βγαίνουν και ενημερώνουν τον εθνικό τύπο για τη συγκεκριμένη θέση που υποστηρίζουν στο Συμβούλιο. Η δε κοινή συνέντευξη τύπου στο τέλος της συνεδρίας του Συμβουλίου συνήθως έχει παρουσία πολύ περιορισμένων, πολύ περιορισμένου αριθμού δημοσιογράφων. Ευχαριστώ πολύ Βιβιάννα. Σε ευχαριστώ για τις δηλώσεις σου, για όλα αυτά τα χρόνια που εργάστηκες ως Επίτροπος μαζί μας. Ξέρουμε ότι έχεις αποφασίσει να σταματήσεις. Όχι, όχι, ως Επίτροπος. Όχι. Μα θα ήσουν υποψήφια για το κοινοβούλιο. Α, όχι, όχι, όχι, όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εγώ είμαι από αυτούς τους επιτρόπους που πάντοτε εκτίθενται στην εκλογική διαδικασία. Πάντοτε. Και πάλι στις εκλογές θα κατεβώ. Και αν πάλι διοριστώ επίτροπος, θα διοριστώ επίτροπος. Εάν δεν διοριστώ επίτροπος, τότε θα στραφώ στο κοινοβούλιο. Αυτή είναι η ζωή. Καλώ λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει τώρα λίγη αυτή η θητεία σου, στο τέλος του χρόνου τουλάχιστον λίγη αυτή η τρέχουσα θητεία και είπες ότι δεν θα είσαι επίτροπο μέσα στην προεκλογική εκστρατεία όπως και ο Μπαρνιάν. Δεν... Λάθος τα κατάλαβα πάλι. Όχι, όχι, όχι. Ω παπα, τι απίθανη παραπληροφόρηση είναι αυτή. Λοιπόν, η συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής δείχνει, λέει, ε, Κοινοβουλίου και Επιτροπής θέλω. λέει ότι μέλη της Επιτροπής μπορεί να κατέβουν στην προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι επίτροποι. Δεν πρέπει να είναι επίτροποι. Πρέπει να πάρουμε δηλαδή άνευ αποδοχών άδεια για την περίοδο της προεκλογικής εκστρατείας. 15 χρόνια άλλωστε αυτό κάνω. Κάθε φορά άνευ αποδοχών άδεια, προεκλογική εκστρατεία και μετά την εκστρατεία ξαναγυρίζω στην Επιτροπή. Και πριν αναλάβει κανείς καθήκοντα ή το αξίωμα καλύτερα του βουλευτή, θα πρέπει να έχει επιλέξει εάν θέλει να είναι βουλευτής ή επίτροπος. Έτσι είναι η κατάσταση. Μάλιστα, για τον Παρόσο ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Γιατί και μετά τις εκλογές κάποιοι επίτροποι δεν εξελέγησαν, δεν, έγιναν, ε, δεν επανεξελέγησαν. Εν πάση περιπτώσει για σένα τέτοιο κίνδυνο δεν υπάρχει. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην περαιτέρω πολιτική σου σταδιοδρομία Ίσως και κάποιοι να σε ακολουθήσουν, ίσως κάποιοι όλοι όχι. Να μην προδικάσουμε τίποτα σήμερα, αλλά ζούμε στον αληθινό και όχι στον ιδεατό κόσμο. Εύχομαι κάθε επιτυχία λοιπόν στις προσπάθειές σου και για όλα αυτά τα οποία έχουμε καταφέρει χαίρομαι πολύ, για τα όσα δεν έχουμε ολοκληρώσει θα δούμε πώς μπορούμε στη συνέχεια με άλλους επιτρόπους και αυτό βέβαια ξέρουμε ότι οφείλεται σε έναν βαθμό στις ε, οικονομικές ε, στα οικονομικά προβλήματα, στα χρήματα που δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε για τα έργα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα για τους συντονιστές έχουμε τίποτα. Όχι, δεν υπάρχουν προβλήματα για τις αποφάσεις των συντονιστών. 14 στα διάφορα. Ούτε εδώ έχουμε τίποτα. Προσεχή συνεδρίαση 12 Φεβρουαρίου. 13 Φεβρουαρίου 9. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και τα ξαναλέμε την επόμενη φορά.